και τώρα ερχόμαστε στην σύντομη παρουσίαση της εξαίσουσης της κυρίας Ρης για τα προβλήματα υγείας που συνδέονται με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δίνω το λόγο στην εισηγήτρια για τέσσερα λεφτά. Ευχαριστώ. Δεν είμαι η πρώτη και προφανώς δεν θα είμαι και η τελευταία η οποία θέλει να καταγγείλει το άρθρο 45 του κανονισμού που περιορίζει τις ε, συζητήσεις, ε, δεν υπάρχει συζήτηση, δεν υπάρχει συνομιλητής για τις ομάδες και θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Γιάλα, την ε, η κυρία Κίνο, τον κύριο Βανίστελ Ρόι και όσους δεν βρίσκονται εδώ και ε, δυστυχώς συζητάμε πολύ σύντομα ε, στις 11 η ώρα το βράδυ ένα θέμα που ενδιαφέρει πολύ τους Ευρωπαίους πολίτες. Το είχαμε αγνοήσει επί 10 χρόνια, δηλαδή σχεδόν ε, ένα αιώνα στις νέες τεχνολογίες για τα Wi-Fi, τα Bluetooth, για τα κινητά τηλέφωνα, ένα σωρό θέματα τα οποία μας περιβάλλουν και μας απασχολούν πολύ και επηρεάζουν πολύ την υγεία μας. Να είμαστε σαφείς σε ένα πολύ ευαίσθητο πλαίσιο χρειάστηκε να εκπονήσω την έκθεση αυτή σχετικά με τους κινδύνους για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία χαμηλής ε, συχνότητος και δίνω ορισμένα παραδείγματα των προτάσεων οι οποίες ελπίζω ότι θα υπερψηφιστούν αύριο την ε, προστασία για τις, τους παιδικούς σταθμούς, τα νοσοκομεία ε, και κατάρτιση μίας διαδικασίας η οποία θα καταστήσει ανεξάρτητη την έρευνα αλλαγή συμπεριφοράς προς το κινητό τηλέφωνο για τα bluetooth για τον περιορισμό της χρήσης στα παιδιά γιατί τις εκστρατείες marketing ε, και ε, για τη συμπεριφορά των, ε, οργαν... των εταιριών κινητής και να υπάρξει ένας περιορισμός του επίπεδου των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που δεν με ακολουθεί σε η Επιτροπή παρόλο που πέρυσι στις 2 Σεπτεμβρίου το ίδιο κείμενο είχε υπερψηφιστεί για ένα για μια άλλη έκθεση ε, σχετικά με τα θέματα υγείας και περιβάλλοντος 2004-2010. Ο στουρθοκαμιλισμός της Επιτροπής δεν συμβάλλει στο να διευκρινιστεί το θέμα για τους Ευρωπαίους πολίτες και οι γνώμες των εμπειρογνωμόνων διαφέρουν. Μία φορά κλείνουν προς ε, τους, ε, τις βιομηχανίες και μία φορά για τους ενδιαφερόμενους Υπάρχουν προτάσεις ε, ε, του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας για να περιοριστεί αυτό το κοκτέιλ των κυμάτων χαμηλής συχνότητος αλλά πιστεύω ότι η λύση δεν είναι η κατάλληλη και ελπίζω ότι δεν θα δούμε στο μέλλον ότι ε, περιπέσαμε σε ε, μια ιστορία η οποία ήταν πολύ επικίνδυνη χρειάζεται ένας ορισμός ο οποίος πρέπει να υπάρξει σήμερα στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και γι' αυτό και η πρόταση των πρασίνων έχει την πλήρη στήριξή μου γιατί ε, συνδυάζεται με την αρχική πρότασή μου να μειωθούν τα επίπεδα εκπομπών που δέχονται οι ε, νέα περιοχές και στην ε, Ουαλονία και στις Βρυξέλλες Βρυξέλλες ε, όπου έχει μειωθεί το επίπεδο. Είμαι η συγκίτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα ήθελα ιδίως ε, να ε, προστατεύσω την έκθεση την οποία έχουμε ψηφίσει στην Επιτροπή και ολοκληρώνοντας έχω δύο μηνύματα. Ο φάκελος αυτός για τις επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων παραμένει ανοιχτός και ελπίζω ότι το επόμενο Κοινοβούλιο το το ξανασυζητήσει διότι η Ευρώπη πρέπει να επανέλθει στη συζήτηση αυτή η οποία αυτή τη στιγμή απλούστατα επιλύεται στα δικαστήρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα θα ακούσουμε τον Επίτροπο Φερχόγγεν. Πρόεδρε, Ευρωβουλευτές, θα ήθελα την Ευρωβουλή και ιδιαίτερα εσάς κυρία Ρίσο, η συγγητρία, να ευχαριστήσω θερμά για αυτή την έκθεση ιδίας πρωτοβουλία για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Πράγματι, πρόκειται για ένα θέμα, τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, που για πολλούς Ευρωπαίους πολίτες ε, είναι ένα πολύ επίμαχο και προβληματικό πεδίο, αλλά πάρα πολύ σημαντικό και για μας εξίσου. Και λόγω του περίπλοκου σύνθετου χαρακτήρα που έχει και λόγω των έντονων αισθημάτων συγκινησιακά που προκαλεί αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερη σημασία με ιδιαίτερα αντικειμενικό τρόπο να συλλέξουμε τα στοιχεία και να τα συγκρίνουμε και να τα αξιολογήσουμε με ιδιαίτερη σύνεση. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς διαρκώς το θέμα και αυτό και μάλιστα βάσει της σύστασης ε, του ε, Συμβουλίου αυτό κάνει. Γι' αυτό σε τακτά διαστήματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις ανεξάρτητες επιστημονικές επιτροπές συλλέγει και ζητεί να υποβάλλονται στοιχεία ώστε σε θέμα πιθανών τέτοιων προβλημάτων σε σχέση με τα ηλεκτρομαγνητικά προβλήμα, ε, παιδεία να είναι πάντα ενήμερη και να γνωρίζει τις εξελίξεις. Η πρόσφατη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιστημονικής επιτροπής ε, εφέτος εγκρίθηκε τον Ιανουάριο 2009 πολύ πρόσφατα. Θα ήθελα να αναφέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις εξελίξεις στα κράτη-μέλη, καθώς επίσης και την ομολογία του 10, καθώς επίσης και των εθνικών δικαστηρίων, όπως για παράδειγμα στη Γαλλία, παρακολουθεί την ομολογία και την εξέλιξή της με ιδιαίτερη προσοχή. Και όσον αφορά και το, τα πεδία ε, έκθεσης ε, των πολιτών σε αυτά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Μπορώ να διασφαλίσω ε, τα μέλη της Ευρωβουλής ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αιτήματα τα οποία περιέχονται σε αυτή την πρόταση ψηφίσματος με ιδιαίτερη προσοχή θα τα εξετάσει. Κάποια στοιχεία να αναφέρω. Πρώτον, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει ήδη ένα πλαίσιο με το οποίο δημιουργούνται τη μέσα για την έκθεση, όρια για την έκθεση σε τέτοιου είδους μαγνητικά πεδία. Δεύτερον, οι μέχρι σήμερα ανεξάρτητες, από ανεξάρτητους επιστήμονες ε, μελέτες την ε, τροποποίηση αυτών των τιμών ε, δεν την δικαιολογούν επιστημονικά και έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί τα επιστημονικά δεδομένα και στοιχεία σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το πεδίο, ώστε να διασφαλίζει αν προσαρμογές των επιπέδων έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι αναγκαίες ή όχι. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι καθήκον της τον διάλογο με τις ε, ανάλογες ε, αντίστοιχες ομάδες που εμπλέκονται σε αυτό το θέμα να τον καλλιεργήσει ώστε με τους πιο σημαντικούς εταίρους να συνεργαστεί ώστε με τον πιο εύθετο ενδεδειγμένο τρόπο να μπορέσει να αντιμετωπίσει και να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στι ανησυχίε των πολιτών. Με ιδιαίτερο τρόπο θέλω να τονίσω ότι και η έρευνα θα πρέπει να συνεισφέρει για την αποσαφήνιση ενδεχόμενων αβεβαιοτήτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Προσπαθήσαμε όπως είδατε και εμείς να μειώσουμε τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία μέσα στην αίθουσα όσο μιλούσα. Σβήστε τα κινητά σας. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Τώρα μένει μια έκθεση της κυρίας Ούρσουλας Γκάτσεκ για τα προβλήματα και προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Το λόγο έχει συγκίτρια για τέσσερα λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πίτρο.